Ζούμε σε μια δημοκρατία και δεν είναι δυνατόν να περιγράφουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ως, δικαστήριο μαριονέτας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλακ δεν είναι εδώ, αλλά σίγουρα θα σημειώσει τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Βάτλη, είστε έτοιμος. Με ναι, συγγνώμη, ξεκίνησα χωρίς να έχω σηκωθεί. Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι γεγονό ότι το δεσμικό αυτό όργανο ενσαρκώνει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Γι' αυτό και πρέπει να πω ότι με κάποια συναισθηματική φόρτιση λαμβάνω το λόγο σήμερα για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την εκπόνηση, την κατάρτιση μάλλον του προπολογισμού για το έτος 2011. Κυρίως γιατί πρόκειται για μια διαδικασία κατάρτιση προπολογισμού λοιπόν για το 2011 βάσει μιας εντελώς νέας διαδικασίας με πολύ σαφώς ενισχυμένο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα εγκαινιάσουμε μαζί λοιπόν αυτή τη ε, διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας για την κατάρτιση του προπολογισμού του 2011. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σήμερα που είμαι εδώ παρόν και ε, εκφωνώ αυτή την ομιλία ενώπιόν σας. Θα ήθελα επίση ε, να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η συνεργασία και αυτή η συζήτηση που θα πρέπει να έχουμε στο πλαίσιο τη νέα αυτή διαδικασία ε, τη Λισαβόνα. Πρέπει να πω ότι είχαμε κάποιες καλές ε, επαφές, οι πρώτοι τριμερείς διάλογοι είχαν καλά αποτελέσματα και αυτό πριονίζεται καλά για το μέλλον. Λυπούμεθα, λέει η Κομισιόν, για την έλλειψη πολιτικής βούλησης κατά την κατάρτιση της θέσης του Συμβουλίου. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή Δημοσιονομική έκανε τη σχετική εργασία. Επιμένω πάντως στο γεγονός ότι η σχετική εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο πολύ σαφών προσανατολισμών που έχει ορίσει στις 16 Μαρτίου του 2010 το Συμβούλιο Κοφίν. Για να σεβαστούμε το πρωτόκολλο 1 για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, εγκρίναμε επισήμως στο Συμβούλιο την θέση μας ε, με τη γραπτή διαδικασία στις 12 Αυγούστου. Δεν ε, στερεί λοιπόν τίποτε αυτό από την πολιτική σημασία ε, για τη διαδικασία κατάρτιση του προβλησμού του 2011. Άλλωστε αποτελεί ε, κάτι καινούργιο για όλους μας με τους νέους αυτούς κανόνες και σίγουρα θα πρέπει να συναγάγουμε τα σχετικά συμπεράσματα για το μέλλον. Όπως είναι προφανές, καταρτίστηκε ο προβλησμός αυτός βάσει ορισμένων αρχών για το σεβασμό των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013. Φυσικά, ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και δεύτερη σημαντική αρχή να εγγυθούμε τα κατάλληλα περιθώρια ώστε διάφορε πολιτικέ θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να μπορούν να διαφανούν ξεκάθαρα και να είναι και αξιόπιστε. Ο προπολογισμό βέβαια καταρτίζεται στο πλαίσιο μια δημοσιονομική λιτότητα. Θα πρέπει να είναι άλλωστε αυτό, γνωρίζουμε ε, ξεκάθαρο και σε όλα τα κράτη-μέλη. Το 2011 θα είναι δύσκολη χρόνια για όλους. Πρέπει λοιπόν και αυτή η δημοσιονομική λιτότητα να είναι εμφανής, να είναι παρούσα και στο σχέδιο προπολογισμού του 2011. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ στις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές ε, του σχεδίου προπολογισμού του 2011 και μετά θα ε, επεκταθώ συγκεκριμένα για κάποιες από τις κατηγορίες προτείνουμε 142 δις ευρώ προπολογισμό ε, σε αναλήψεις ε, πληρωμών. ...778 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει και ένα, μια προσαρμογή με 3,6 δις ε, σε ό,τι αφορά σαν λήψη υποχρεώσεων σε σχέση με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή μείωση κατά της τάξης του 2,8%. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο επίσης έλαβε υπόψη ε, τις δείξεις που το έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πληρωμή των προγραμμάτων 2007-2013 της πολιτικής συνοχής και ιδίως λάβαμε υπόψη τις τελευταίες πληροφορίες ε, για ε, την ταχύτητα εκτέλεσης των μεγάλων μιζώνων σχεδίων. Βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση ορισμένων σχεδίων. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι μετά τη μία του Συμβουλίου, το σύνολο των ψώσεων πληρωμών ε, εξακολουθεί να αυξάνει σημαντικά, κατά 2,91 δηλαδή, σε σχέση με το 2010. 1% λοιπόν ε, περισσότερο σχεδόν από τη μηδενική αύξηση. Πληθωρισμός δηλαδή που έχει οριστεί στο το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και στη μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις τελευταίες δημοσιονομικές προβλέψεις ε, για τα σύνολα πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων που αυξάνονται σημαντικά και στην απόλυτη αξία τους ε, και σε ποσοστά. Δεν πρόκειται να επισέλθω στην κάθε κατηγορία του προπλήσμου ξεχωριστά. Απλά να σα υπενθυμίσω στην κατηγορία 1α γνωρίζουμε ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πολιτική για την νεολαία είναι προτεραιότητα. Αυτό άλλωστε ε, αναγράφεται και σε όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγματι ε, είναι λίγο χαμηλότερε οι προτάσει μα σε σχέση με αυτέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ο προπολογισμό αυτό είναι σαφώ αυξημένο σε σχέση με το προπολογισμό του 2010. Σε ό,τι αφορά το 1β, εδώ πραγματικά το σύνολο των ποσών ε, του προπολογισμού αυτού καθορίστηκαν πραγματικά με βάση την τρέχουσα εκτέλεσή τους. Ε, έχουμε σεβαστεί αυστηρά την εκτέλεση όπως την βλέπουμε σήμερα να υπενθυμίσω για την ε, κατηγορία 4, για το τίτλο 4, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις οικονομικές, κοινωνικέ προκλήσεις ε, και σε διεθνέ επίπεδο κυρίω. Και είμαστε, έχουμε την επίγνωση ότι νέε δημοσιονομικέ προκλήσει ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και για τον προπολισμό υπερθμών 5 δεν τροποποιήσαμε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια για το δικαιωτικό του προπολογισμό. Νομίζουμε όμως ε, ότι κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες να παραμείνει εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, δείχνοντας έτσι ότι κάθε θεσμικό όργανο καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες ε, προκειμένου να σεβαστούμε τον ε, οδικό χάρτη που έχουμε σήμερα. Για να ολοκληρώσω, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτή τη παρουσίαση ήταν πολύ σημαντικό να είναι εδώ παρόν το Συμβούλιο για να σα παρουσιάσει τη λογική, τη συλλογιστική που ακολουθήσαμε για την κατάρτιση του προπολογισμού. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσω αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα ε, σε σχέση με τη θέση που έχει οθετήσει το Συμβούλιο. Ωστόσο, αυτό που περιμένω είναι οι διαπραγματεύσει μα με το Κοινοβούλιο να είναι επικοδομητικέ ε, και να καρποφορήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή της ε, στη διάρκεια της διαδικασίας που σίγουρα θα είναι γεμάτη προκλήσεις. Δεν μπορώ όμως να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου χωρίς να αναφέρω το budget review που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του μήνα αυτού. Οι προτεραιότητες για τον προπολογισμό του 2011 και συγκεκριμένα στρατηγική 2020 χωρίς ε, καμία αφιβολία θα είναι η προτεραιότητά μας για τα μελλοντικά έτη. Σε αυτή λοιπόν ε, την οπτική γωνία ήδη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αρχίσει να εξετάζει σε βάθος ε, την χρηματοδότηση και τη διάρθρωση του Και θέλω να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία θα φροντίσει να δώσει το Συμβούλιο ιδιαίτερη προσοχή στο budget review, στην αναθεώρηση του προπολογισμού. Για να επανέλθω τώρα στον προπολογισμό του 2011, αυτόν καθεαυτόν, πρέπει να σα πω ότι η, Ευρωπαϊκή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια τα οποία θα συναντήσει στη διαδικασία αυτή. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα διαπραγματευτούμε τις διατάξεις, με βάση τι διατάξει τη της Λισαβόνα και ελπίζω πραγματικά να καταφέρουμε να δείξουμε ότι αυτή η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη διαδικασία θα στεφθεί με επιτυχία. Δεν ε, θα αφιστούμε προσπαθειών ω Συμβούλιο ώστε ο προπολογισμό μα ε, να ωφελήσει έναν ω τον το μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, φορολογουμένων δηλαδή, από του οποίου άλλωστε εξαρτάται και η χρηματοδότηση του προπολογισμού μα. Ευχαριστώ. Thank you. And now for the commission, Mr. Lewandowski. Ο κύριος Λεβαντόφσκι, εκ μέρους της Κύριε Πρόεδρε, Είμαστε τώρα στην κρίσιμη φάση της αιτήσεως διαδικασίας αλλά δεν είναι μια διαδικασία ρουτίνας, γιατί για πρώτη φορά εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και φτάνει τώρα η κρίσιμη στιγμή για τον προπολογισμό. Στον τελευταίο τριμερή διάλογο δεν συμφωνήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, δεν είχαμε μεγάλη πρόοδο, αλλά τουλάχιστον αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής για το 2010. Επομένως τώρα έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του Συμβουλίου και πρέπει να λάβει θέση το Κοινοβούλιο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και θα συνεχίσει η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τι διαδικασίε και στα δύο σκέλη τη Δημοσιονομική Αρχή του Προπολογισμού. Όμω, ε, είναι επίση πολύ σημαντικό ότι έχουμε ακόμη και ένα ολόκληρο πακέτο ε, ε, μέτρων προσαρμογή σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και απαιτείται λοιπόν καλή θέληση και από τι δύο πλευρέ για να συμφωνήσουν. Αυτό το οποίο τώρα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον Νοέμβριο είναι ένα ευρύ φάσμα δύσκολων θεμάτων προς επίλυση. Ένα πολυδιάστατο λοιπόν πακέτο συνδιαλλαγής για τον Νοέμβριο. Όσον αφορά τα θέματα ουσίας, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, ε, υπάρχουν κάποιες περικοπές πληρωμών κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο προϋπολογισμού, γνώριζε τα προβλήματα και τα μέτρα λιτότητα στα κράτη-μέλη ε, και γι' αυτό συντάξαμε τον προϋπολογισμό 4 δισεκατομμύρια ευρώ πιο κάτω από την οροφή της δημοσιονομικής προοπτικής. Και επιπλέον όλες τις αυξήσεις, κύριε Υπουργέ, τις ε, συγκεντρώσαμε στην κατηγορία 1 σε θέματα τα οποία οδηγούν σε νέες θέσεις απασχόλησης και ήταν, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σαν ένα μικρό πακέτο ενίσχυσης της απασχόλησης. 96% των αυξήσεων βρίσκονται στην κατηγορία 1 ως μέτρο που αποδεικνύει την ευθύνη που αναλαμβάνουμε και η συνοχή κινείται τώρα πλέον με την σωστή ταχύτητα στο μέσο της περίοδου εφαρμογής των προγραμμάτων, ενώ στην αρχή κινείται πιο ε, αργά. Ε, μιλάμε και για μέτρα ε, μείωσης δαπανών στα προενταξιακά μέτρα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε σε σχέση με την κατανομή κονδυλίων μεταξύ χωρών θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρός ε, ε, για τα διοικητικά ε, θέματα. Αυτό το οποίο περικόπτεται είναι οι γραμμές διοικητικής υποστήριξης. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχουν σχέση και με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα και στη φυσική καταστροφή στο Πακιστάν και για την ανθρωπιστική βοήθεια και ε, για την επίγουσα βοήθεια. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή την περασμένη εβδομάδα, αλλά αυτό απαιτεί ε, ε, κόστος διαχείρισης. Υπάρχει και κάτι άλλο που ήταν επίσης αντικείμενο περικοπών για τα executive agencies και για την ε, έρευνα που διαχειρίζονται το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτά αυξάνεται και πρέπει να αυξηθούν κατά ένα δισεκατομμύριο το 2011. Η Επίμετρον θα ήθελα να ζητήσω και από τα δύο σκέλη της Δημοσιονομικής Αρχής να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά τις ανησυχίες αυτές που εξέφρασα όταν θα διαπραγματευτούν την τελική συμφωνία που θα είναι πολυδιάστατη για το 2011 και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε θα προσπαθήσουμε ε, να παίζουμε το ρόλο του ενδιάμεσου με τρόπο επικοδομητικό πάντοτε για να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα για το 2011. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Η κυρία Γεωτζερεύσκα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο προπολογισμό του 2011 δεν είναι ο μόνος ο οποίος καλύπτεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα, όπως είπατε άλλωστε, αλλά είναι ουσιαστικά ο πρώτος προπολογισμό στα πλαίσια του οποίου εφαρμόζονται οι νέε πολιτικές, οι οποίες εμπνέονται από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Είναι ο πέμπτος προϋπολογισμός των δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2013 και σε αυτή τη φάση έχουμε μάθει πολλά θα έλεγα για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των δημοσιονομικών πρακτικών μας μέχρι τώρα. Ευχαριστώ την Βελγική Προεδρία για τις προσπάθειες της, αλλά ανησυχώ γιατί υπάρχουν 7 κρατημέλη που έχουν καταψηφίσει την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο. Έχω την αίσθηση ότι όταν οι Υπουργοί Οικονομικών από τις χώρες εξετάζουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς και βλέπουν το σκέλος της συνεισφοράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο το οποίο κάνουν είναι να σκέφτονται το πώς θα περιορίσουν τη συνεισφορά τους, χωρίς να σκέφτονται τι γίνονται τα χρήματα τα οποία δίδουν και ποιες θα είναι οι συνέπειες της μείωσης αυτή της συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να σταματήσει από πλευρά των διαφόρων υπουργών. Λυπάμαι επίσης γιατί το Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει μέχρι τώρα και προχωρά σε μειώσεις του προϋπολογισμού σε συγκεκριμένες γραμμές. Ελπίζω στο μέλλον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί στο Συμβούλιο έχουν αυτή την περιοριστική πρακτική. Η διαδικασία η δημοσιονομική πρέπει να είναι όσο περισσότερο ανοιχτή γίνεται και όσο περισσότερο λεπτομερής γίνεται. Πρέπει λοιπόν οι προτάσεις που κάνουμε για τις συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού να μην αφορούν μόνο αυστηρά λογιστικές ανησυχίες, αλλά την ουσία των πολιτικών προς τις οποίες στοχεύουν. Λοιπόν, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εκπλήσουν κανένα, αφορούν ε, την νεότητα, αφορούν την κινητικότητα των εργαζομένων, αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όταν το Συμβούλιο λοιπόν προτείνει τέτοιες σημαντικές περικοπές στις βασικές αυτές προτεραιότητες και αναφέρομαι στα προγράμματα της διαβίου κατάρτισης, τότε τι είδους διάλογο κάνουμε με το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι στα πλαίσια της επόμενης διαδικασίας συνδιαλλαγής να μπορέσουν τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν με το Συμβούλιο, γιατί αλλιώς οι δυσκολίες θα είναι τεράστιες, αν όχι αξεπέραστες. Δεν πρέπει να προχωρούν σε τέτοιου είδους προτάσεις για μειώσεις. Εμείς προετοιμάζουμε τώρα τη δική μας ανάγνωση, έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία και ελπίζουμε να υιοθετήσουμε τη θέση μας μέχρι το τέλος του μήνα και ελπίζω ότι στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου να έχουμε κλείσει τη διαδικασία και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας να υιοθετήσουμε ένα καλό προϋπολογισμό, ένα επικοδομητικό προϋπολογισμό σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία. κυρία Τρούπελ, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε του Συμβουλίου, κύριε εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, κ. Λεβαντόφσκι, αγαπητοί συνάδελφοι. Γνωρίζουμε ε, πως ε, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολιτικοί ζούμε μέσα σε κλίμα πολιτικής λιτότητας και πώς τα κράτη-μέλη επιθυμούν να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Θέλουμε να φροντίσουμε την ισοσκέληση του προϋπολογισμού και σε πνεύμα δικαίου προς τις επόμενες γενναίες και ούτως ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες να ασκούμε την πολιτική μας διαφορετικά ε, πνιγόμαστε εμείς οι ίδιοι ως πολιτικοί αν δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους και το απαραίτητο περιβάλλον. Αυτό απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη αλλά θα ήθελα ε, να μιλήσω γιατί δεν είμαστε όλοι στην, σε ταυτόσιμη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δημιουργήσει χρέη, είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται και από τη συνθήκη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, και αυτό είναι κάτι που θέλησαν τα κράτη-μέλη, με τη συνθήκη της Λισαβόνας απέκτησε νέα καθήκοντα, νέες αρμοδιότητες που πρέπει να διεξαχθούν και στην Επιτροπή και στην ε, πολιτική ενέργεια και στην εξωτερική πολιτική και σε τομεί και θα πρέπει να είμαστε σε θέση τα νέα αυτά καθήκοντα τα οποία μας δόθηκαν από τη συνθήκη να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όπως αρμόζει. Ω εισηγήτρια ε, θέλω να πω ότι απαιτείται η σωστή ισορροπία μεταξύ των νέων αρμοδιοτήτων και παράλληλα μια υπεύθυνη πολιτική προϋπολογισμού και πολιτική δαπανών, πράγμα το οποίο δεν έχει εξευρεθεί ακόμη. Για όλες τις νέες θέσεις ε, για τη διοίκηση έχει ε, αρνηθεί την συμφωνία του Συμβούλιο για το ελεκτικό συνέδριο, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά όχι για το ίδιο το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι άδικο, γιατί σε πιο μικρά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα να εργαστούν σωστά. Και αν θέλουμε σωστό έλεγχο από το Ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει να δώσουμε στους συνεργάτες μας, στους συναδέλφους μας αυτά τα όργανα να μπορούν να ταξιδέψουν, να μπορούν να έχουν περισσότερο προσωπικό και να ανταποκριθούν στο έργο του. Και αυτή η σωστή ισορροπία νομίζω ότι είναι σημαντικό πολιτικό πολιτικό καθήκον και είναι και ένα σημαντικό μήνυμα που θα δώσουμε και προ τα κράτη-μέλη και προ του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο με εκπλήσει επίση είναι το κόστο για τη διεύρυνση μειώνονται οι πόροι από το Συμβούλιο, αλλά δεν έχει αλλάξει η ημερομηνία προσχώρησης. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει στην πράξη κάτι τέτοιο. Επίσης, αν θέλουμε σωστό προϋπολογισμό, θα πρέπει να είμαστε ε, σωστά προετοιμασμένοι και να μην έχουμε περικοπές σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, ε, ε, υπάρχει το πρόγραμμα της ατομικής ενέργειας, το οποίο επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να περικοπεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουκ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε πρόσωπο του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Οι συγκητέ ήδη έδωσαν μια αξιολόγηση τη θέση του Συμβουλίου και εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο εκ μέρου τη Επιτροπή. Θα ήθελα εξ αρχή να πω ότι είμαι πεπισμένη ότι η Προεδρία του Συμβουλίου από πλευρά Βελγίου κάνει τη δουλειά τη όσο μπορεί καλύτερα. Μπορεί να κάνει τη δουλειά τη όμω τόσο καλά όσο τις επιτρέπει το σύνολο του Συμβουλίου. Και δυστυχώ εδώ πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι κακό. Το Συμβούλιο, ως συνήθως, δεν θυμάμαι τίποτα διαφορετικό εξάλλου, ε, κόβει από την πρόταση της Επιτροπής, από το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής και στις πιστώσεις υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Και γι' αυτό και αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Αυτό το κάνει το Συμβούλιο παντού. Δεν προσπάθησε το Συμβούλιο να δει πού θα είχε νόημα να κάνει περικοπές και πού όχι. Το αποτέλεσμα είναι 780 εκατομμύρια λιγότερο στις υποχρεώσεις και 3,6 δις λιγότερα στις πληρωμές. Και αν το δούμε αυτά, αυτό στην πράξη, αν δούμε, δούμε τι πλήττεται από αυτές τις περικοπές και πάλι βλέπουμε ε, τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο δημιουργήσαμε από κοινού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από κοινού συμμετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις διαφορετικά αυτοί οι οργανισμοί δεν θα υπήρχαν, δεν θα είχαν δει το φως. Τώρα όμως αν δεν τους διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά για την οποία τους δημιουργήσαμε, τη δουλειά που τους αναθέσαμε, θα έπρεπε να τους κλείσουμε αυτούς τους οργανισμούς κάθε ευρώ προ την κατεύθυνση αυτή θα ήταν τί δαπάνη, θα ήταν σπατάλη αν δεν χρειαζόμαστε αυτού του οργανισμού. Μετά υπάρχει το θέμα του Executive Agency που ασχολείται με την εφαρμογή του πολιετούς προγράμματος. Αν δεν διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους, το πρόγραμμα είναι νεκρό. Αυτό θέλουμε. Κάποιοι από το Συμβούλιο θεωρούν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερες προσπάθειες ε, για να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Αλλά στη διαδικασία του προϋπολογισμού περικόπτονται ακριβώς αυτά τα τμήματα του προϋπολογισμού που θα έπρεπε να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ε, ανταγωνιστικότητα, κατηγορία 1α. Το ίδιο και για, τι για τις πολιτικές. Γίνονται περικοπές ακριβώς ε, εκεί όπου χρειαζόμαστε πόρους, μείον ένα δισεκατομμύριο. Δεν είναι λογικά όλα αυτά και δεν είναι και καθόλου έξυπνα. Θέλουμε με πολιτική υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε τον προϋπολογισμό και μάλιστα ουσιαστικά. Για να μπορέσει η Ευρώπη να έχει μια προστιθέμενη αξία για όλους τους πολίτες, ούτως ώστε να είναι και ουσιαστικό αυτό το οποίο κάνουμε και να το βλέπουν οι πολίτες. Έτσι θα θέλαμε να είναι ο εταίρος μας στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Και ας δώσουμε στο, προς το παρόν τουλάχιστον τον τελευταίο λόγο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. σχετικά με την έλλειψη της δυνατότητας συζήτησης για το σύνολο των γραμμών του προϋπολογισμού όπως είχε προταθεί από το Συμβούλιο. Εγώ νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές θα γίνουν σε κάποια φάση. Ε, οφείλουμε να τις κάνουμε. Είναι συζητήσεις για τις προτεραιότητες ε, οι οποίες θα χαρακτηρίσουν τον προϋπολογισμό του 2011. Αλλά είναι σαφές επίσης ότι η συμφωνία δεν ήταν εύκολη στο Συμβούλιο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και θα πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός σε επίπεδο Συμβουλίου έγινε αντικείμενο ψηφοφορίας, του οποίου την έκφαση δεν γνωρίζαμε και αυτό οφείλεται στη δημοσιονομική κατάσταση την οποία γνωρίζει κάθε χώρα στο εσωτερικό της. Μια οικονομική κατάσταση δύσκολη και μια δημοσιονομική κατάσταση δύσκολη. Παρά όμω τις δυσκολίες αυτές, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε στις χώρες μας αντίστοιχα, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010 έχει αυξηθεί. Αυτή η αύξηση του 2,91%. Το λέω αυτό για να κλείσω ότι πολλοί θα ήθελαν το ποσοστό αυτό να είναι μεγαλύτερο, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2010. Η κυρία Χάουγκ υπογράμμισε το 1β του προϋπολογισμού. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το 1β σε σχέση με το 2010 αυξάνεται κατά 14%. 14%. Το να λέμε λοιπόν ότι δεν έχει λάβει υπόψη το Συμβούλιο τα ειδικά χαρακτηριστικά του 1β ενώ το αυξάνει κατά 14% είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι το Συμβούλιο αναγνωρίζει το θέμα και αυτή η αναγνώριση δεν έχει παρατηρηθεί σωστά από, τους, από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Να πω επίσης στους εισηγητές για το 2011 ότι στα πλαίσια της παρέμβασής μου θελήσαμε να υπογραμμίσουμε την προσπάθεια που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφερθήκατε και στο 1-1 το οποίο υπογραμμίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ υπογράμμισα στην παρέμβασή μου ότι το Συμβούλιο πράγματι θέλησε να δείξει ότι στα πλαίσια της προσπάθειας την οποία κάνει υπάρχει η επιθυμία να βρεθεί μια συμφωνία ιδιαίτερα στον τομέα της νεότητας. Και υπάρχει ένα άνοιγμα στον τομέα αυτής της πολιτικής ακριβώς γιατί το έχει ζητήσει ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν μία από τις βασικές του προτεραιότητες. Θα ήθελα να επιθυμίσω επίσης ότι στο κεφάλαιο 5 και στο θεσμικό κομμάτι είναι σαφές ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες. Είναι επίσης αλήθεια, στα πλαίσια του προϋπολογισμού που παρουσιάζει το Συμβούλιο, ότι δεν έχουμε θίξει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως έχει. Νομίζω όμως ότι έχει σημασία κάθε θεσμικό όργανο να κάνει κάποια μορφή εξοικονόμησης, κόστους και όλοι να δείξουμε το παράδειγμα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η τόσο δύσκολη δημοσιονομικά χρονιά για να κλείσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουν και άλλες συναντήσεις, καρποφόρες ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω να είναι καρποφόρες όπως είπα, έτσι ώστε ο προπολογισμό για το 2011 να κλείσει γρήγορα. Να υπενθυμίσω ότι ο προπολογισμό αυτός δεν είναι ένας εύκολος προπολογισμό. γιατί έχουμε νέες διαδικασίες, γιατί έχουμε νέες πολιτικές τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε και επίσης γιατί δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την δημοσιονομική κατάσταση, την δύσκολη στην οποία βρίσκονται όλες οι χώρες μέλη. Το σύνολο των δημοσιονομικών στόχων τους οποίους θα πρέπει να πετύχουμε θα το κάνουμε αυτό συνειδητοποιώντας τις δυσκολίες αυτές. Και ελπίζω από κοινού να καταλήξουμε σε μια δημοσιονομική λύση αποδεκτή για το 2011 και να μπορέσουμε από κοινού να δείξουμε ότι αυτή η νέα της διαδικασίας που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας θα στεφθεί από επιτυχία, από έναν προϋπολογισμό δηλαδή, στον οποίο όλοι θα συμφωνήσουμε. Thank all. That now closed. Σας ευχαριστώ όλους. Πέρας του συγκεκριμένου θέματος. Περνάμε τώρα στο χρόνο ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Αλλά στις 8.30